εγκρίνονται αυτές, ε, ε, αυτοί οι διορισμοί. Επίσης, ε, με χαρά θα χαιρετήσω επίσημα, στα, επίσημα θεωρία τον κύριο Κομπάκιτζε που είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας καθώς και την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει. Ils effectuent ce jour une visite. Πρόκειται για μια επίσκεψη εργασία στο Ευρωκοινοβούλιο και μα τιμούν με την παρουσία του ε, στη διάρκεια τη συζήτηση και τη ψηφοφορία. Σήμερα σα καλωσορίζουμε θερμά και περνάμε στι ψηφοφορίε. Ξεκινάμε με την έκθεση του κυρίου Τάκουλα. Πρόκειται για μια μόνο ψηφοφορία με ονομαστική κλίση.